Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε παρακαλώ το ταχύτερο, καθώς στις 9 πρέπει να ε, αποχωρήσουμε από την αίθουσα, γιατί έχει έκτακτη συνεδρίαση και η Επιτροπή Απασχόλησης στη συνέχεια. Γερμανικά τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην σημερινή έκτακτη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο. Χαίρομαι που παρά την πολύ πρωινή ώρα μας προήρθατε πολύ άριθμοι. έχω εγκρίνουμε την ημέρη σε διάταξη, ελπίζω. Την Τρίτη με το email σας ενημερώσαμε ότι είχαμε τη γνωμοδότηση για το, για, για το Invest EU για την τρίτη αφήση. Γιατί η αρμόδια καθήλυνη επιτροπή πρόκειται να ε, διεξαγάγει την ψηφοφορία της αργότερα, οπότε και εμείς δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να εγκρίνουμε την πρόταση της ημερήσιας διάταξης όπως έχει, αν δεν έχετε αντίρρηση την εγκρίνουμε. Ανακοινώσεις της Προέδρου δύο μόνο. Διερμηνία στις εξής γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, εσθονικά, ουγγρικά, πολωνικά και ρουμανικά. Και για άλλη μια φορά υπενθυμίζω ότι μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου αυτή η συνεδρίαση. Και έτσι περνώ στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Δύο είναι οι ψηφοφορίες που έχουμε σήμερα για, για νομοθετικές γνωμοδοτήσεις. Ξεκινώ με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με εισηγήτρια την υποφαινομένη. 228 τροπολογίες λάβαμε. Ευχαριστώ όλους τους και ηγητές. Ήταν καλές και επικοδομητικές οι συνθήκες μας στις οποίες εγκρίναμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Σε πολλά σημεία μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και με την υποστήριξη της συναδέλφου Σόιντροβα από την Επιτροπή Απασχόληση πιστεύω μπορούμε να εξασφαλίσουμε συμπερίληψη και των τροπολογιών μας στην Επιτροπή ΕΜΠΛ. Σε κάποια σημεία θα χρειαστεί παραπάνω προσπάθεια, γιατί δεν είμαστε απόλυτο ικανοποιημένοι από όλε τι ε, προόδου. Χρειάζεται παραπάνω δουλειά και για να συμπεριληφθούν αυτέ τι τροπολογίε στην έκθεση τη ΕΜΠΛΗ. Και έτσι προχωρώ στην, τροπο... στην ψηφοφορία. 138 και 139 ταυτόσημες. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Θα σας παρακαλέσω όμως να σηκώνετε το χεράκι, αλλιώς δεν βλέπω ε, υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθησαν. 140 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη. 141, 142 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Πέρας. 12 υπέρ 11 κατά εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όχι, όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Έπρεπε να έχω περάσει ήδη στην συμβαστική υπαριθμόν 1. Συμβαστική 1 λοιπόν υπέρ κατά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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 198 έχει αποσυρθεί. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, ξαναρχίζω. Τη 200 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 209 υπέρ κατά αποχές Ας το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ, 10 κατά, απερίφθη, 210 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη 211 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 213 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 και 24 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 219 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε τη 219 Αρχιτεί ψηφοφορία Πέρας Εγκρίνεται 15 υπέρ 10 κατά 220 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 221, 222 μαζί υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 223, 224 ταυτόσημες υπέρ, κατά αποχές απερίφθησαν 225 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 226 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 227 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 231 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 233 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 234 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 237 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 238 έχει αποσυρθεί 239 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 230, 240 έχει αποσυρθεί 241 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 200 Ζητώ συγγνώμη, γυρνώ. Λάθος σας τα διάβασα. Τη 240 πρέπει να την ψηφίσουμε. Η 240 παρακαλώ, υπέρ, κατά. Αποχέ απερίφθη. Και τώρα πάμε στη 242. 242 υπέρ, κατά. Αποχέ απερίφθη. 243 υπέρ, κατά. Αποχέ απερίφθη. 244 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 245 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 250 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 251 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 252 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 253 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 255 256 υπέρ κατά αποχές απερίφθησαν 257 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 32 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 35 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική, ε, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 80 και 82 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 103 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 104 και 105 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απερίφθησαν συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 ελέγχουμε την 123 μάλλον πρώτα αρχίζουμε έλεγχος 123 πέρασε εγκρίνεται 17 υπέρ 9 κατά 10 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130-131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 28 συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 137 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συνολική ψηφοφορία ονομαστικά παρακαλώ για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία geschlossen 18 υπέρ, μία ψήφος κατά, 6 αποχές, μεγάλη η πλειοψηφία ε, με την οποία εγκρίνεται η έκθεση. Ευχαριστώ θερμά και ελπίζουμε αυτές τις ευφύες μας τοποθετήσεις να τις υιοθετήσει και η Επιτροπή ΕΜΠΛ. Και προχωρώ στην ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Πέθρου και τα με τον κύριο Στρογεύσκη, εισηγητή, είναι παρόν. Θες να πεις κάτι, θέλετε να πείτε κάτι, όχι. Πάμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 47 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 48 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 49 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 50 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 52 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 53 έχει αποσυρθεί 54 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 93 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Ας επαληθεύσουμε αν θέλετε. Πέρας. 17 κατά. 8 ψηφί. Πέρα περίφθη. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθει. 96 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 99 έχει αποσυρθεί 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 102 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 103 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά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 Απερίφθη 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 29 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 30 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 34 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 ναι, ναι, ναι, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται... Να σας πρόχνω λίγο σε Ή να σου δώσω ένα ε, να υποστηρίζει το χέρι σου. 40, 40 ε, λοιπόν υπέρ κατά υπέρ. Ε, εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται και έτσι τελική ψηφοφορία ονομαστικά παρακαλώ. Geschlossen. Πέρας. 20 υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές. Και εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ταχύτατε οι συνομιλίες και οι εργασίες μας. Τώρα μπορούμε να παραδώσουμε την αίθουσα στην ΕΜΠΛ. Η προσεχή μας συνεδρίαση είναι τη Δευτέρα με την Διακοινοβουλευτική Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα συνεδριάσουμε μαζί με τη δική μας την Επιτροπή. Παρακαλώ να είμαστε πολύ άριθμοι παρόντες. Το ίδιο και για το πρωί της 20ης Νοεμβρίου όπου έχουμε την Ολομέλεια. Το δε απόγευμα έχουμε την τακτική μας συνεδρίαση. Με τα συνήθι θέματα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και θα σας δω τη Δευτέρα. Η Σίλβια. Ε, ε, μόνο, μόνο κάτι. Ξέρω ότι η Προεδρία έδωσε μεγάλη μάχη με την Προεδρία του Κοινοβουλίου για να έχουμε τις ε, μεταφράσεις στις διάφορες γλώσσες στα, στα πάνελ. Αυτό όμως δεν ε, ε, επέτραπη και είναι πολύ σοβαρό γιατί εμείς βρισκόμαστε σε μεγάλη δυσκολία το να καλούμε τα εθνικά κοινοβούλια και να μην μεταφράζουν τα κείμενα δεν είναι ένα καλό δείγμα. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, θα ήθελα να το υπογραμμίσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί η διάσκεψη των Προέδρων δεν δέχτηκε κάτι τέτοιο. Θα το πούμε υπεύθυνα στο τους το ότι ζητάμε την κατανόησή τους, αλλά ήθελα να το αναφέρω διότι δεν είναι καλή εικόνα για τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες όλοι. Η Πρόεδρος, ναι, όντως κατέβαλα πολλές προσπάθειες και μάλιστα προσπάθησα να πείσω και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, όπως στείλαμε στις διάφορες συναφείς ε, ε, υπηρεσίες πολυάριθμες επιστολές. Η απάντηση ήταν πάντα ότι α, είναι πολλές οι συνεδριάσεις που ταυτόχρονα λαμβάνουν χώρα και οι που δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η διερμηνία. Τουλάχιστον για τα δύο, α, το ένα από τα πάνελ έχουμε διερμηνία τη Δευτέρα. Ελπίζουμε μέχρι τη Δευτέρα κάτι να γίνει, αν και δεν έχω προσδοκίες. Θα ήταν καταστροφικό βεβαίως κάτι τέτοιο, γιατί στο κύριο αυτό, ε, στην κύρια αυτή εκδήλωση που αφορά το, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς με παρουσία Ευρωπα... Εθνικών Κοινοβουλίων να μην υπάρχει διερμηνία θα είναι καταστροφή. Είναι κάτι βεβαίως το οποίο δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων να είναι σε θέση να μιλήσουν αγγλικά ε, και να καταλάβουν επομένως είναι καταστροφή για μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε πει ότι ματαιώνουμε την πρώτη μέρα. Αλλά θα ήταν ακόμα χειρότερο. Και γι' αυτό και δεν την ε, ματαιώσαμε. Σαμπίνε Φερχάιεν. Ναι, πρέπει να πω ότι η διοίκηση του Κοινοβουλίου έχει φερθεί κατά κάποιο απαράδεκτο θα πω τρόπο. Δεν μπορεί να μου πει ότι είναι μία τακτική συνεδρίαση πιο σημαντική από αυτή τη συνεδρία στη δική μας, γιατί είναι καθήκον μας τακτικό να έχουμε την επικοινωνία με τα εθνικά κοινοβούλια και έχει ε, ανεβάσει σε ψηλό μπαϊράκι την, ε, το έτος Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς στο Κοινοβούλιο, στην προβολή του. Πάνω από, λοιπόν, πάνω από όλα λοιπόν αυτό η πολυγλωσία δεν είναι πολιτιστική κληρονομιά. Έχουν κρατήσει κόσμο σε επιφυλακή για να τον διαθέσουν αν χρειαστεί να γίνει καμιά συνομιλία για το Brexit που δεν θα γίνει. Οποιοςδήποτε λοιπόν έχει η αδίποτε πρόσβαση σε οποιονδήποτε εδώ μέσα στο κοινοβούλιο, από τη διοίκηση, από οτιδήποτε και μπορέσουμε να δείξουμε, είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να δείξουμε ξεκάθαρα ότι ο αγώνας μας είναι για την πολυγλωσία εδώ μέσα και εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού δεν πρέπει να δεχόμαστε στο έτος πολιτιστικής κληρονομιάς να κάνουμε συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια χωρίς διερμηνία. Είναι απαράδεκτο. ας μας πούνε ότι κάνουν οικονομία ε, στα χρήματα και έτσι θα τα κάνουν όλα στα αγγλικά, αλλά όχι στη συγκεκριμένη συνεδρία. Τι λες, να ματαιώσουμε την πρώτη μέρα δηλαδή, κύριε Φερχάιεν. Όχι. Αυτό που προτείνω είναι να προσπαθήσουμε όλοι με όποιες γνωριμίες έχουμε τρόπους επικοινωνίας κτλ. Επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να έρθει το θέμα όχι μόνο σε επίπεδο επιτροπής μας, αλλά σε ανώτερο επίπεδο πολιτικό να ασκηθεί πίεση, διάσκεψη των Προέδρων. Μήπως μια από τις τακτικές επιτροπές μπορεί να τα καταφέρει μόνο στα αγγλικά. Αντί για μας. Καλώς ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άλλη μια φορά. Διατυπώνουμε εμεί τι άλλο τη δυσφορία μας γιατί είναι σκανδαλώδες το... Σκανδαλώδα ή τα τεκτενόμενα. Αυτά λοιπόν. Ε, θα εύχομαι πάντως. Καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε τη Δευτέρα.